προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την έχει υποβάλει ο κύριος ε, Πάρης εκ μέρους της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου και η ερώτηση αυτή αφορά την μεσογειακή δίαιτα. Και τώρα, από και τον ε, λόγο, για πέντε λεπτά ο κύριος Πάρης για να παρουσιάσει την προφορική του ερώτηση. Πρόεδρε, Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί θεωρείτε τόσο καλή την μεσογειακή δίαιτα, την εφαρμόζετε και την θεωρείτε ιδιαίτερα θετική. Σαν πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας είχαμε πολλά, είχα πολλά πράγματα να συζητήσω. Τη μία φορά συζητήσαμε για τη μεταφορά των ζώων που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και τώρα μιλάμε για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που είναι η μεσογειακή δίαιτα. <laughs> αυτό είναι ένα από τα καθήκοντα τα οποία έχω αναλάβει ως πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και στις 16 Ιουλίου πέρυσι στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε την πλήρη υποστήριξή της για τον, για τον χαρακτηρισμό της μεσογειακής δίαιτας σαν μνημείο της παγκόσμιας άιλης κληρονομιάς της UNESCO. Η υποψηφιότητα θα εξεταστεί το 2009 από την αρμόδια δια επιτροπή της UNESCO. Και θα ήθελα να ρωτήσω, προτίθεται η Επιτροπή να καταρτήσει συγκεκριμένη και συντονισμένη στρατηγική για να υποστηρίξει αυτή την υποψηφιότητα, διότι προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα. και εκπροσωπώ την Επιτροπή Γεωργίας εδώ, αλλά νομίζω ότι εκπροσωπώ και όλα τα μέλη όταν μιλάμε για την δίαιτα, διότι ένα από τα σημαντικά πράγματα της Ευρώπης είναι η ποικιλία και η διαφορετικότητα, ε, η πολιτισμική. Και μία από τις πολιτισμικές διαφορές ε, που μας χαρακτηρίζει είναι το φαγητό. Τώρα θα μου πείτε τι είναι μια μεσογειακή δίαιτα και νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε αρκετά για αυτό το θέμα σήμερα το πρωί, αλλά είναι μια δίαιτα όπου ε, ε, παίζουν σημαντικό ρόλο το ελαιόλαδο, τα ψάρια, ε, τα φρούτα, τα λαχανικά και όπως βλέπετε και από το μέγεθός μου την υποστηρίζω πλήρως. Βέβαια είναι μια υγιεινή δίαιτα διότι είναι μια πολύ καλή πηγή για τα καλά λιπαρά, για τα, για τα προωθεί την ε, υγεία και βλέπουμε ότι οι προ, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να, ε, προ, να προλάβει και κάποιες ε, ψυχικές ή πνευματικές διαταραχές. Όσοι όσοι έχουμε πάει στις μεσογειακές χώρες ψάχνοντας για ήλιο βρίσκουμε και πολύ καλό φαγητό και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά σε έναν κόσμο όπου συνεχώς βλέπουμε ότι τα πάντα γίνονται ομοιόμορφα. Βλέπουμε ότι η νέα γενιά ε, βομβαρδίζεται από αλυσίδες fast food, δεν πρόκειται να τις αναφέρω όλες εδώ σήμερα, αλλά βλέπουμε ότι όλες αυτές οι αλυσίδες ε, έχουν εγκατασταθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ναι, το fast food έχει μια θέση, Απ' την άλλη πλευρά όμως ήταν τραγικό εάν τα επόμενα χρόνια ταξίδευες, ταξιδεύεις σε όλη την Ευρώπη και το μόνο που συναντάς είναι fast φουντάδικα. Το βλέπουμε αυτό και σε πολλές χώρες, σε πολλές πολιτείες της Ηνωμένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στις δυτικές ακτές παραδείγματος χάρη, όπου δεν μπορεί να βρει τίποτα άλλο τόσο από φασφουντάδικα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το αποφύγουμε στην Ευρώπη. Επομένως πρέπει να υποστηρίξουμε τη μεσογειακή δίαιτα και είναι πολύ καλό για την πολυπολιτισμική, για πολιτισμική μας ε, ε, διαφορά. Ε, και αυτό το οποίο ήθελα να πω σήμερα το πρωί είναι ότι εγώ υποστηρίζω πλήρως ε, τη μεσογειακή δίαιτα, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν ε, εμφανίζομαι εδώ μπροστά σας σαν πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας υποστηρίζοντας μόνο τη μεσογειακή δίαιτα, διότι υπάρχουν και άλλες δίαιτες στην Ευρώπη που είναι εξίσου καλές αλλά με διαφορετικές αξίες αν θέλετε. Ε, λοιπόν, θα ήθελα πραγματικά να μου πει η Κομισιόν τι προτίθεται να κάνει για να υποστηρίξει αυτή την ε, πρωτοβουλία. Διότι μιλάμε για, την, ε, για μνημείο της παγκόσμιας άλλης κληρονομιάς. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, προς τον κύριο Πάρης. Και τώρα ο Επίτροπος και ο Σπίτιλα θα απαντήσει εκ μέρους της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Πρώτα, πρώτα θέλω και εγώ να σας τονίσω ότι είναι πολύ σημαντική η υγιεινή διατροφή για την πρόληψη των ασθενειών. Γνωρίζετε ότι έχουμε τη Λευκή Βίβλο που φύγει τα προβλήματα της υγείας που προέρχονται από κακή διατροφή ε, και για τη κατάσταση που κάποιος είναι υπέρβαρος ε, του Μαΐου του 2007 εμείς που συνεχώς προσπαθούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την βελτίωση της ε, διατροφής και την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Είναι θέματα επομένως δημόσιας υγείας, διατροφής, μεταφορών, περιφερειακής επιτροπής, <clears throat> αθλητισμού λαμβάνουμε υπόψη και τις στατιστικές αλλά φυσικά και κυρίως τη γεωργική πολιτική και άρα σας ε, τονίζω ότι είχαμε μια πρωτοβουλία αναλάβει που αφορούσε την ε, διανομή φρούτων στα σχολεία. Με το πρόγραμμα εκείνο θέλαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να κάνουν ένα σωστό ξεκίνημα στη ζωή τους. Αυτό ξεκίνησε την σχολή περίοδο 2009-2010 9 ε, εκατομμύρια ευρώ διαθέσαμε για να υπάρξει μεταφορά και διανομή φρούτων στα σχολεία. Ε, τώρα για το ερώτημα ακριβώ που μου υποβάλλατε για την ε, ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής ως άιλης πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO ο προκάτοχός μου ο κύριος Κυπριανού στο Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2007 είχε φέρει προς το θέμα αυτό. Εμείς χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία εκείνη και βεβαίως ε, θέλουμε να υπάρχει γενή διατροφή σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Πάντως η Επιτροπή δεν έχει τις ε, αρμοδιότητες ούτως ώστε να προβάλλει στην UNESCO αυτό το αίτημα. Δεν είμαστε ως Κομισιόν μέλος της UNESCO. Δεν μπορούμε να εμπλακούμε σε μια τέτοια ε, απόφαση εκ μέρους της UNESCO. Πάντως θα θέλαμε τα κράτη-μέλη να το καταφέρουν. Και ε, επομένω θα τους υποστηρίξουμε πλήρως. Και τώρα έχουμε τους αγορητές των ευρωπαϊκών, των, συγγνώμη, των πολιτικών ομάδων. Πρώτα-πρώτα για τρία λεπτά η κυρία Μιγγέλα για τους σοσιαλιστές. Πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας όσον αφορά αυτή την υποψηφιότητα που θέλουμε να υποστηρίξουμε στην UNESCO για τη Μεσογειακή Δίαιτα. Άκουσα την απόφαση του κυρίου Επίτροπου, άρα θα πρέπει να καταλάβετε εδώ πρόκειται για ένα πολιτιστικό αγαθό. έχουμε το θέμα της διατροφής που είναι κάτι ευρύτερο από ένα απλό πρότυπο. Ε, άρα αυτό θα πρέπει να το λάβετε υπόψη γιατί αυτό αφορά την υγιεινή ζωή, αφορά επίσης και την πρόληψη των ασθενειών που έρχεται όταν κανείς δεν διατρέφεται σωστά, όταν δεν ε, ασκείται. Όμως, εδώ έχουμε κάτι ευρύτερο, έχουμε ένα ολόκληρο τρόπο ζωής, χαρακτηριστικό το, το, το, τη σχέση του κανείς με, με, με το με το, με το να μοιράζεται την τροφή με παρέα. Αφορά το, ακόμα και την ύπεθρο, αφορά το τοπίο. Ε, μιλάμε για διαδρομή αιώνων που κατέληξε να, να γίνει μια ολόκληρη τέχνη. Υπάρχουν γιορτές, υπάρχει ολόκληρη κουλτούρα σε σχέση και γύρω από την ε, μεσογειακή δίαιτα. Και για μένα την ίδια αλλά και για άλλους ε, αυτό πάει να πει η Μεσογειακή Ιδιαίτα και γι' αυτό και προωθούμε αυτή την υποψηφιότητα βεβαίως και συμφωνούμε με την ε, θετική στάση της Κομισιόν και φυσικά έχετε δίκιο ότι στην UNESCO δεν είσαστε μέλος της Κομισιόν ξέρουμε ότι δεν ε, συμμετέχετε στην διαδικασία λήψης εκείνων των αποφάσεων όμως μπορείτε να βοηθήσετε αυτή την υποψηφιότητα με κάποιο είδους ε, έμεσους τρόπους και έτσι να υπάρχει υποδοχή θετική αυτής της ε, πρότασης και άρα έτσι μπορείτε να εμπλακείτε σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσατε να κάνετε και κάποια επίσημη δήλωση όσον αφορά αυτή την υποψηφιότητα. Να υποστηρίξετε την υποψηφιότητα Έχουμε και άλλους φορείς διεθνείς, την Οργάνωση για την Υγεία, τη ΦΑΟ ε, και ε, οπότε από όλες αυτές τις οπτικές γωνίες θα μπορείς να δει το θέμα για να βοηθήσει. Άρα μπορείτε να συμμετάσχετε σε κάποιες τέτοιες συγκεκριμένες κινήσεις υπερκρατικού χαρακτήρα. Άλλωστε μιλάμε τώρα για την χρονιά του διαπολιτισμικού διάλογου. Και άλλωστε η πρόταση για την ζωική διατροφή ε, θα γίνει σε συνεργασία και με την γείτονά μας χώρα το Μαρόκο. Και έτσι θα προωθήσουμε τρόπο ζωής και διατροφή που να είναι υγιεινά. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να γίνουν διπλωματικές κινήσεις. Να ληφθεί υπόψη φυσικά ο σεβασμός που οφείλουμε προς τις τρίτες μεσογειακές χώρες που δεν είναι στην Ένωση και έτσι, Επίτροπε, μπορείτε να βοηθήσετε και να αποδείξετε το πόσο θετικά βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία για όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίους μήνες. Και τώρα, για τους φιλεύθερους δημοκράτες θα λέει το ρόλο ο κύριος Χατζημαρκάκης. Δύο λεπτά. Ευχαριστούμε, Νίλ Πάρης, για την ερώτηση. Ευχαριστούμε και την Κομισιόν για την απάντηση. Πολλά πράγματα ζηλεύουν στην Ευρώπη, την Ευρώπη να τον κόσμο, για το πώς ζούμε, για τα συστήματα κοινωνικής μας ασφάλισης και επιπλέον και για την διατροφή μας. Και βεβαίως ε, αυτή ανήκει και η πιο υγιεινή από όλες, η μεσογειακή διατροφή. Και βεβαίως εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι κατά κύριο λόγο μιλάμε για διατροφή της Κρήτης, μεγάλων Νομάτων της Ελλάδας και της Νότιας Ιταλίας. Και χαρακτηριστικό στατικό αυτής της διατροφής είναι το ελαιόλαδο. Ένας λόγος παραπάνω, κύριε Σπίτλα, και απευθύνουμε σε ολόκληρη την Κομισιόν, να προστατεύσετε αυτό το αρχαίγωνο ευρωπαϊκό προϊόν. Και βεβαίως φρούτα, λαχανικά, χαιρετίζουμε το ότι προσφέρονται φρούτα και στα σχολεία προγραμματικών, προγραμματικό ψάρια και κρασί. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο τε... κάτι το οποίο δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal το Σεπτέμβριο του 2008 πως όλα αυτά συνεισφέρουν στο να μειώσουν τις ε, καρδιοσθένειες, το διαβήτη τύπου 2, μια, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή επιδημία, τον καρκίνο και όλα αυτά τα προλαμβάνουν και μειώνουν και τις ε, επιδράσεις του. Κάτι το οποίο θα δείτε σε οποιοδήποτε νεκροταφείο της Κρήτη, από την οποία κατάγεται και ο πατέρα μου. Βλέπετε τη μεγάλη ηλικία των ανθρώπων, σε τη μεγάλη ηλικία πεθαίνουν. Και γεγονός είναι βεβαίως πως ε, η δίαιτα αυτή κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για τις προσπάθειες αυτές. Αλλά πρέπει να δούμε πως εάν η Κίνα και η Ινδία ακολουθήσουν τον αμερικανικό τρόπο διατροφής έχουμε τρία αρνητικά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα η υγεία τους βεβαίως θα γίνει χειρότερη. Δεύτερον θα οδηγηθούμε σε μαζική κτηνοτροφία με ό,τι σημαίνει αυτό για το περιβάλλον. Και τρίτον βεβαίως θα έχουμε και επιπτώσει για το κλίμα γιατί το κρέας αυτό θα είναι κατά κύριο λόγο βοδινό και γνωρίζετε πως τα βοηδοί παράγουν μεθάνιο. Αυτά σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Πάρης. Μέτσι. Κύριος Μουζουμέκη για την Ευρώπη των Εθνών για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της μεσογειακής δίαιτας η οποία προτείνεται να γίνει άλλο μνημείο ανθρωπότητας από την UNESCO μας υπενθυμίζει ε, τι σημασία έχει αυτή για χώρες που προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, το Μαρόκο αλλά αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί εκεί πιστεύω ότι πρέπει να ξαναφτιάξουμε τον δεσμό ο οποίος έχει αποδυναμωθεί μεταξύ της παραγωγής και αυτού που εμφανίζεται κάθε φορά στο τραπέζι μας. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κόσμο το ρητό νους υγιής ενσώματι υγιή με φαγητά, με τροφές που είναι φυσικές, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά η, κοινότητα έχει η επιστημονική κοινότητα έχει συγκεντρώσει πολλά στοιχεία για το τι ε, ευνοεί την υγεία μας. Ας πούμε το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, το ε, κρασί, τα πορτοκάλια της ε, Σικελίας που είναι αντιοξυδοτικά. Ελπίζω τον στόχο αυτό να τον συμμερίζονται και άλλες χώρες της Μεσογείου, που χρειάζεται ωστόσο μια ειδική στρατηγική που μόνο η Επιτροπή μπορεί να ερμηνεύσει και να καθοδηγήσει. Ευχαριστώ για δύο λεπτά εξ ονόματος της ΓΚΟΕ, της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ο κύριος Γκερέιρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να προωθήσουν και να διαφυλάξουν τις, ε, τη λαϊκή κουλτούρα, ιδιαίτερα στον τομέα της διατροφής, όπως ε, για παράδειγμα η υποψηφιότητα της μεσογειακής δίαιτας στην UNESCO ως ε, κληρονομιάς τη νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Ε, ο στόχος θα μπορούσε να είναι να γίνει ε, πιο γνωστή μια δίαιτα που ανήκει στους που γνωρίζουν οι λαοί της Μεσογείου και που επιδοκιμάζουν όλοι οι ειδικοί. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η δίαιτα περιλαμβάνει παραδοσιακά τρόφιμα της Μεσογείου, ε, ξηρούς καρπούς, λάδι, ε, ε, ε πρόβιο, κρέας, οποροκυπευτικά, ψάρι. Ωστόσο, η μείωση, βλέπουμε μείωση του πληθυσμού που ακολουθεί την δίαιτα αυτή με συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να προωθηθεί η παραδοσιακή μεσογειακή δίαιτα, ιδιαίτερα στα πλαίσια της κοινή γεωργικής και της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Μέτρα που αφορούν την γεωργία, ε, την οικογενειακή γεωργία και την αλληλεία στη Μεσόγειο εξασφαλίζοντας τα έσοδα των ε, αλλιέων και των καλλιεργητών. Κάτι που θα, θα δυναμώσει και την ε, τοπική αγορά. Ζητούμε να υπάρξουν μέτρα που θα προστατεύουν τον πληθυσμό, τον τοπικό πληθυσμό που γνωρίζουν την παραγωγή και τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων αυτών. Πρόκειται για μέτρα που πρέπει να λάβει κυρίως η Επιτροπή. Μπαίνουμε στους αγορητές, των, ε, τους ατομικούς αγορητές. Καταρχάς, ο κύριος Κάπουλα Σάντο για δύο λεπτά πρώτα. Μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν είναι πολύ εύκολο να χειριστεί κανείς ένα τέτοιο θέμα που συνδυάζει τρία βασικά θέματα, την υγεία, τον πολιτισμό και την οικονομία. Η μεσογειακή δίαιτα θα συγκεντρώνει και αυτά, έχει, συγκεντρώνει και τις τρεις αυτές διαστάσεις. Από υγείας δεν υπάρχει καμία επιστημονική αμφιβολία για τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής δίαιτας που στηρίζονται σε νοπά προϊόντα όπως τα τοπικά δημητριακά, το ρύζι, τους ξηρούς καρπούς, την τοπική, τα τοπικά οποροκυπευτικά, τα προϊόντα της θάλασσας και το ελαιόλαδο και το κρασί. Από άποψη πολιτισμού, η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων αυτών συνεχίζουν πανάρχιες παραδόσεις των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων μέθοδοι που εξακολουθούν σήμερα να χρησιμοποιούνται στην περιοχή της Μεσογείου. Όσον αφορά την οικονομική διάσταση, ο τομέας της ε, γεωργίας, της αλληλείας και του αγροτοτουρισμού που εμπλέκονται στη μεσογειακή δίαιτα μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου, κάτι που πρέπει να ενισχυθεί. Κυρίως όσον αφορά τη γεωργία. Η μεσογειακή γεωργία είναι ανταγωνιστική γεωργία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να εξακολουθεί να επωφελείται από τα μέτρα της αγροτικής πολιτικής. Θα πρέπει επίσης να συγχαρούμε τις Ισπανικές αρχές που κατάφεραν να πείσουν την UNESCO να αναγνωρίσει την ε, ε, μεσογειακή δίαιτα ως στοιχείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό κάτι, είναι κάτι που πρέπει να υποστηριχθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι ενδιαφέρει μόνο στις μεσογειακές χώρες αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ένα λεπτό για τον κύριο Ταταρέλα. Πρόεδρε Επίτροπε, η παχυσαρκία γίνεται ένα σοβαρό βαρύ, μεγάλο πρόβλημα για όλη την Ευρώπη, ιδίω για τους νέους. Με βάση τους ειδικού, αν θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών μας, πρέπει σε καθημερινή βάση να ε, επιστρέφουμε στις παραδόσεις της μεσογειακής διατροφής, που είναι η μόνη εξασφάλιση για τη ζωή που καμιά οικονομική κρίση δεν θα μπορέσει να θίξει. Η έρευνα του κ. Καρίνο, γνωστού Ιταλού ΣΕΦ και μια ολόκληρη επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την, ε, ε, που έκανε έρευνα για την μεσογειακή δίαιτα και ζήτησε να υιοθετηθεί ως ε, κοινή κληρονομιά τη της ανθρωπότητας φέρνει πίσω την κουζίνα στις αρχές της ποιότητας. Η μεσογειακή κουζίνα δεν είναι ψωμί και ζυμαρικά, είναι και φυσικό στυλ και τρόπο ζωής. Η μεσογειακή δίαιτα περνά από το καλό κρασί, από το ε, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και από την ε, αντιμετώπιση της φύσης ως κομμάτι της ζωής. Χάρη στην μεσογειακή δίαιτα, οι Ιταλοί έχουν είναι η, εθνότητα με το με, μεγαλύτερο μέσο όρο ζωή στην Ευρώπη και ε, να κλείσω λέγοντας ότι η γερουσία της Ιταλίας ε, υιοθέτησε πρόσφατα ομόφωνα ένα κείμενο που αναγνωρίζει τη μεσογειακή διέτα ως κληρονομιά της ανθρωπότητας. Εύχομαι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει την ίδια άποψη και να, και να προσαρμοστεί σχετικά η Επιτροπή. Συγγνώμη. Πόσο χρόνο έχω πρόεδρε, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, επίτροπε, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, ε, ευγνωμονώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του Κοινοβουλίου του κύριο Πάρης, που προώθησε την προφορική αυτή ερώτηση μετά την σημαντική ακρόση των εμπειρογνωμόνων που διεξαγάγαμε στην Επιτροπή αυτή στο παρελθόν. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η μεσογειακή διατροφή αποτελεί τμήμα της ε, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Επίρου μας, όπως αδιαμφισβήτητο είναι ότι στηρίζεται και έχει αποτέλεσμα θετικό για την υγεία. Το εντοπίζει αυτό και η ίδια η λευκή βίβλος της Επιτροπής για την παχυσαρκία, θεωρώντας ότι η μεσογειακή δίαιτα είναι ένα ιδιαίτερα κατάλληλο φυσικό φάρμακο. Τα πλονεκτήματα στην υγεία αποδεικνύονται επιστημονικά και είναι πολύ ευνοϊκά δεκτά και στο εξωτερικό, ξεκινώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σημαντικό λοιπόν να διευρυνθεί η έννοια χωρίς να ε, αποδυναμώνεται η πρωτοτυπία τους. Γι' αυτό η αναγνώριση της μεσογειακής δίαιτας από την UNESCO καθορίζει και κατοχυρώνει το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό της ε, δίαιτας της Μεσογείου. Και με τον όρο ιδιαιτερότητα σήμερα εννοώ τη μεσογειακή διατροφή αλλά όχι ως ε, μόνο ε, αυτό το, δεν είναι μόνο αυτό το χαρακτηριστικό, το ίδιο το χαρακτηριστικό της ε, μεσογειακής διατροφής. Κύριε Επίτροπε, εσείς δεσμευτήκατε όπως και ο, και ο προκάτοχός σας να θεωρείτε ε, σημαντική την πρωτοβουλία αυτή και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Υπογραμμίσατε ότι η Επιτροπή δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για τα θέματα UNESCO, ωστόσο πιστεύω ότι θα μπορούσατε να λάβετε θέση, να προχωρήσετε, διακόπτεται ο μιλητής. Ο κύριος Μπατιλόκιο, για ένα λεπτό. Ξεκινάμε, πρόεδρε, από την έννοια. Πολλές μελέτες λένε ότι η μεσογειακή δίαιτα μειώνει την παχυσαρκία και τις καρδιοπάθειες, βελτιώνει την ανθρώπινη υγεία σε πολλές πτυχές. Ωστόσο, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να επιβάλλουμε τη μεσογειακή δίαιτα σε όλους, ούτε να ε, την ενθαρρύνουμε σε σχέση με άλλες μορφές διατροφής που μπορεί να προσαρμόζονται καλύτερα σε διαφορετικές περιοχές και διαφορετικά κλίματα. Ε, ωστόσο, πρέπει να προστατεύσουμε την δίαιτα αυτή και τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό για να αποφύγουμε εξωτερικές παρεμβάσεις που θα επιδεινώσουν και θα μειώσουν την, την θα επιδεινώσουν τη θα μειώσουν την αξία της. Θα πρέπει όπως και άλλες πολιτισμικές ε, εκφράσεις των Ευρωπαίων να προωθηθεί και να, και να υποστηριχθεί. Ένα μοντέλο, πρόκειται για ένα μοντέλο που μιμείται ο υπόλοιπος κόσμος. Καλό είναι λοιπόν να διαφυλάξουμε τις ιδιαιτερότητές της για να αποφύγουμε ένα καθαρά ευρωπαϊκό στοιχείο κληρονομιάς να χαθεί μεταξύ των κόσμων. Ευχαριστώ. Μπαίνουμε τώρα στην ε, διαδικασία των, ε, του Catch the Eye. Ο κύριος Ικέσκη έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η μεσογειακή δίαιτα βεβαίω αξίζει να προστατευτεί και να προωθηθεί για πολλούς ε, λόγους. Είναι κάτι το οποίο είναι δημοφιλές και ταυτόχρονα έχει και όφελος ε, για την υγεία, κάτι το οποίο είναι σημαντικό για όλες τις γενιές, τους νέους ηλικιωμένους και τους ε, μεσήλικες. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες και δεδομένα και ευρήματα που έχουν συσσωρευτεί που αποτελούν καλή βάση για να αξιολογήσουμε και να υπερασπιστούμε την μεσογειακή δίαιτα. Τα πλεονεκτήματα για την υγεία είναι σαφή, ωφελεί η δίαιτα στα καρδιαγιακά νοσήματα και είναι κάτι που όλοι θα έπρεπε να απολαμβάνουμε. Ο κύριος Ματσάκης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η δίαιτα είναι γνωστό ότι επηρεάζει την υγεία και είναι πλέον αδιαμφισβήτητο τη μεσογειακή δίαιτα επί τη βάση των παραδοσιακών διατηρητικών συνθήκων της Νότιας Ευρώπης όπως η Κύπρος και η Κρήτη οδηγεί σε μακροβιότητα και υγεία ενώ η αμερικανική ε, διατροφή, το junk food δηλαδή, τα hamburger, οι πατάτες τηγανιτές ε, κλπ οδηγούν σε μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολύ περισσότερα ως Κομισιόν για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τη μεσογειακή δίαιτα στα σχολεία και απαγορεύεται η δίαιτα που, θα, που έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί η βλάβη στην υγεία. Κύριε Επίτροπε, δεν καταλαβαίνω πρέπει να σας πω για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέλος της UNESCO. Μήπως θα έπρεπε να γίνει. Κύριε Τομασέφσκα. Panie Przewodniczący, Κύριε Πρόεδρε, είναι βεβαίω καλύτερο το να έχει κανείς ε, καλή διατροφή και να μην ε, υποφέρει η υγεία του από το να αντιγράφει τις ε, μόδες ε, της ε, διατροφής. Βεβαίως το να μειώσουμε την ε, χολυστερίνη είναι κάτι που θα μας ωφελήσει όλους και ακόμη καλύτερο το να βασιζόμαστε σε μακροχρόνιες παραδόσεις που ακριβώς αυτό μας προσφέρει η μεσογειακή δίαιτα. Και χαίρομαι που θα προσθεθεί στην παγκόσμια κληρονομιά μέσω της UNESCO. Περαιούται τώρα η συζήτηση με την παρέμβαση του, του συνονόματου μου κ. Μαρτίνες, Γάλλου συνονόματου. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που είναι ένας Βρετανός, ο συνάδελφος Πάρης που υπέβαλε το κείμενο αυτό. Πολύ καλά έκαναν οι Ρωμαίοι που πήγαν στη Μεγάλη Βρετανία και πέρασαν όλα αυτά, το κρασί ας πούμε. Συμβολικά λοιπόν θα πρέπει το θέμα της διατροφής να προωθηθεί και δεν είναι παρά θα πρέπει η Κομισιόν να αποκαταστήσει τις ενισχύσεις στα προϊόντα και να, κάνει, να επανορθώσει αυτά που έχουν συμβεί κατά το, του ελαιολάδου, των ελαιοδέντρων σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατά τις ε, των, του κόκκινου τόνου και ε, της... Ε, συμπεριφοράς που έχει επιφυλαχθεί στα αμπέλια τα οποία εκριζώνονται και βεβαίως ε, ε, τα ίδια συμβαίνουν στην Πορτογαλία με το ε, κατσικίσιο τυρί κλπ. Λοιπόν. Το λόγο έχει για να ολοκληρώσει συζήτηση ο κύριος Σπίντλα. Επίτροπος κύριος Σπίντλα. Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την στρατηγική που δημοσιεύεται στην Λευκή Βιβλίο υποστηρίζει όλες τις προτάσεις, τις στάσεις που οδηγούν σε υγιεινή ε, διατροφή. Στηρίζει ενεργά όλες αυτές τις πρωτοβουλίες η Κομισιόν αλλά δεν ε, μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τόσο περιορισμένη και συγκεκριμένη ε, δίαιτα καθώς υπάρχουν τεράστιες ε, διαφορές μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών και διαφορές μεταξύ μεμονωμένων ε, μεσογειακών κρατών. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως αυτό το οποίο δήλωσα στα εισαγωγικά μου σχόλια, δηλαδή πως η Κομισιόν υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία συμπερίληψης της μεσογειακής δίαιτας στην πολιτική κληρονομιά της UNESCO. Ε, δεν το υποστηρίζουμε. Οπωσδήποτε το υποστηρίζουμε. Παρά το ότι δεν ε, είμαστε μέλος της UNESCO υπάρχουν τρόποι να στηρίξουμε αυτή την υποψηφιότητα. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω μία παρέμβαση με την οποία διαφωνώ. Εγώ δεν βλέπω κάποιον λόγο για να επανεξετάσουμε την έδρα της σχετικής κοινωνικής υπηρεσίας η οποία είναι αυτή τη στιγμή στην Φιλανδία. Δεν ε, φαντάζομαι πως όσοι ε, εργάζονται για αυτή την υπηρεσία δεν είναι ικανοί να εκπληρώσουν την ε, εντολή που έχουν λάβει. Θεωρώ πως η έδρα αυτή επελέγει σωστά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ τον Επίτροπο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ κρατών ή ομάδων. Πάντως σίγουρα στην συζήτηση που είχαμε εδώ σήμερα δεν διαπιστώθηκαν διαφορές. Δεν υπήρχαν αποκλήσεις ε, από τη Γερμανία και την Πολωνία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο από τη μια μεριά, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κύπρο από την άλλη. Νομίζω ότι εκφράστηκε εκτίμηση με ομοφωνία προς την πρωτοβουλία αυτή και υποστήριξη προς την πρωτοβουλία αυτή. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Θα διακόψουμε για λίγα λεπτά. Τελειώσαμε την συζήτηση νωρίτερα και γαλήνια ούτως ώστε να ακούσουμε όλους κάτι που αποτελεί καλό ξεκίνημα του νέου έτους και της ολομέλειάς μας κατά το νέο έτος. Στις 12 λοιπόν θα ξαναρχίσουμε για τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ.